Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ εκείνου του βουλευτέ οι οποίοι συνυπέγραψαν αυτή την ε, δήλωση. Στην Ολομέλεια τη 17η Δεκεμβρίου του 2009 το Κοινοβούλιο είχε καταθέσει μια, ε, μια, ένα αίτημα προς την ε, νομική του επιτροπή για την, άρση της ασυλίας, για, το, για την εξέταση άρση ασυλίας του ενός βουλευτή και δόθηκε η απάντηση ότι σε θέματα ε, πολωνικής ασυλίας θεωρείται ότι δεν είναι η νομοθεσία δεν επιτρέπει η νομοθεσία την ε, κατάθεση ενός τέτοιου αιτήματο. Με βάση την πολωνική νομοθεσία. Επίσης υπάρχει μια πρόταση για τον Γιώχαν Κορνέλιους Ντεν ε, ως ε, μέλους της Επιτροπής για τη Συνεργασία με τις ΗΠΑ. ευχαριστώ τον κύριο Πλάνη, σε ρωτώ αν υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτό.